Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μια γνωστοποίηση. Στη Δευτέρα της 3 Απριλίου, Απριλίου ε, βάσει του άρθρου γάμα του κανονισμού ε, έγιναν κάποιες ε, δηλώσεις για τη διοργανική ε, συμφωνία βάσει του κανονισμού 69 παράγραφος 1. Τώρα θα